Ε, Καλώ ήρθατε όλοι. Ξέρω πώ είναι λίγο νωρί. Ε, καλώς ορίσατε. Ωστόσο, χαίρομαι που σα βλέπω όλου εδώ. προ ενημέρωσή σας, σήμερα όλε οι συνεδριάσει καλύπτονται από τι 23 γλώσσε τη Ένωση. Εάν βάλετε λοιπόν τα ακουστικά σα, μπορείτε να διαλέξετε ποια γλώσσα θέλετε να ακούσετε και μάλιστα σα παροτρύνουμε να το κάνετε, καθώ και να μιλήσετε στη γλώσσα σα αργότερα, ώστε να πάρετε μια πραγματική γεύση του τι σημαίνει να είστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να ακούς και να μιλάς στις 23 γλώσσες που μιλούνται εδώ και να μπορείς να καταλάβεις και τους ομιλητές που μιλάνε ε, βέβαια στη γλώσσα σας. Εγώ λέγομαι Χριστίνα, είμαι εδώ ως ε, συντονίστρια της ε, πρωινής αυτής συνεδρίασης, της προθέρμανσης. Θα κάνουμε μια σύντομη και ελπίζω και... Ε, ε, ενημερωτική και συναρπαστική συνεδρίαση τώρα. Πριν να αρχίσουμε τις επόμενες δύο συνεδριάσεις θα είναι ο διάλογος των πολιτών με τον Επίτροπο και την απογευματινή συνεδρίαση που ε, αφορά το σώμα αλληλεγγύης. Γι' αυτό θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω τον συντονιστή που θα αναλάβει αργότερα, τον Κριστόφ. Τίνα. Yes. Ε, ευχαριστώ πολύ Χριστίνα. Πολύ ωραία είναι που σα βλέπω όλου εδώ. όπω είπε και η Χριστίνα, εγώ θα συντονίσω τη δεύτερη συνεδρίαση με τον Επίτροπο Ναύρατζιτ, όπου θα έχετε εσεί την ευκαιρία να συνομιλήσετε άμεσα με τον Επίτροπο. Θα ακούσει τι απόψει σα, τι ερωτήσει σα. Πραγματικά προσβλέπω στον ε, διάλογο που θα γίνει σε λίγο και τώρα σα αφήνω στα καλά χέρια τη συναδέλφου μου Χριστίνας. Θα τα πούμε αργότερα. Σας ευχαριστώ και πριν να βουτήξουμε στα βαθιά, στα, στα ουσιαστικά θέματα, θα δώσουμε το λόγο στον Ζαν Μαντούκ, που είναι ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, σε αυτές τις εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια στιγμή ένας τύπος με γραβάτα παίρνει το λόγο. Σήμερα αυτό είμαι εγώ. Αλλά μην φοβάστε, δύο λεπτά μόνο θα μιλήσω και αυτό κυρίως επειδή θέλω επισήμως να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτό το δημοκρατικό θεσμό σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή 23 μέρες πριν από τις ε, επόμενες ευρωεκλογές. Είμαστε πολύ ευτυχείς που είστε όλοι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια, ε, από, από την Ευρωβουλή η Ευρωπαϊκή Ομάδα των Νέων. Γιατί όπως σας είπα Είμαστε λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογέ. Το θέμα της συζήτηση και των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα είναι η δημοκρατία και εγώ. Και Καλύτερο μέρος για να συζητήσει κανείς για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από ότι το ημικύκλιο της Ευρωβουλής. Ακριβώς αυτό είναι ο χώρος, το, η αίθουσα όπου ε, δύο-τρεις μήνες από τώρα θα είναι γεμάτη από τους καινούριους ευρωβουλευτές που κατά τη διάρκεια των επομένων πέντε ετών θα σχηματίσουν το μέλλον της Ένωσης, θα αποφασίσουν για τους νέους κανόνες, νέους νόμους, για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει, θα προοδεύσει ή όχι τους πέντε, τα επόμενα πέντε χρόνια. Και αυτό θα εξαρτηθεί και από εσά, από τι δικέ σα ψήφους που θα ψηφίσετε στι 26 ε, Μαΐου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συζήτηση και η σημερινή εβδομάδα σημαντικό είναι να συμμετέχετε σε όλα τα σεμινάρια και τι δραστηριότητε. Είναι πολύ σημαντικό που έχετε τη δυνατότητα να ανταλλάξετε απόψει με ανθρώπου που προέρχονται από τι διάφορε χώρε, αλλά τελικά νομίζω ότι το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε ώστε να εξασφαλίσετε ότι εσεί θα αποφασίσετε σε τι είδου Ευρώπη που θα ζήσετε τα επόμενα χρόνια και να μην αποφασίσουν οι παλιότερες γενιές που αποφασίζουν ε, κατά κάποιο τρόπο μέχρι τώρα για, το, για τη ζωή σας και το μέλλον σας. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να μην ξεχάσετε και να πάτε να ψηφίσετε και αυτό είναι και το μήνυμα που περνά στις οθόνες του ημικυκλίου. Ότι δηλαδή θέλουμε να ενθαρρύνουμε εσά, αλλά και εσείς τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους συναδέλφους σας, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν ότι, να εξασφαλίσετε ότι το μέλλον θα αποφασιστεί από εσά και όχι από κάποιον άλλον. Είμαι πραγματικά ευτυχής που είχατε την ευκαιρία να έρθετε στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Είναι ενδιαφέροντες καιροί, συναρπαστικοί καιροί, αλλά δεν είναι όλα ξεκάθαρα μπροστά μας. Αναλάβετε λοιπόν την ευθύνη σας ε, να πάρετε πολύ στα σοβαρά τις επόμενες ευρωεκλογές γιατί αφορούν εσάς και το μέλλον σας. Και πάλι σας ευχαριστώ και να περάσετε καλά αυτή τη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Ζερμέν. Ε, this time voting. Όπως ακούσατε λοιπόν ήδη, αυτή τη φορά εγώ και οι φίλοι μου ψηφίζουμε. Αυτός ο τίτλος πώς προέκυψε. Τον Φεβρουάριο ε, ξεκινήσαμε ένα διαγωνισμό στο Facebook ζητώντας σχέδια δράσης από όλους τους νέους που ενδιαφέρονταν να μας προτείνουν δηλαδή πρόγραμμα σχέδιο για τις ευρωεκλογές για να πείσουμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Και ανάμεσα σε όλους συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Επιλέξαμε τρεις νικητές, οι οποίοι είναι σήμερα εδώ μάλιστα, κάθονται εδώ στην πρώτη σειρά. Και θα τους δώσουμε το λόγο θα μας παρουσιάσουν γρήγορα γρήγορα τις προτάσεις τους ε, αυτές που κέρδισαν δηλαδή, που ήταν οι πιο καινοτόμες ή ολοκληρωμένες προτάσεις για το τι μπορεί να κάνει κανείς και ο καθένας θα έχει δύο λεπτά για να παρουσιάσει την πρότασή του, να δώσει κάποια έμπνευση για το τι μπορεί να γίνει από τον καθέναν από εμά. Γιατί αυτή τη φορά η προεκλογική εκστρατεία δεν είναι μόνο θεσμικό θέμα, είναι κάτι που όλοι μας ε, στο οποίο όλοι μας μπορούμε να συμμετέχουμε. είναι λοιπόν ο Ευάγγελος Κάσος, συνοικητής από την Ελλάδα, ο Χαβιέ Ροντρίγκε από την Ισπανία και ο Ντόμα Κόσκοβατς. Και θα σας δώσω λοιπόν το λόγο στον έναν μετά από τον άλλον με αυτή τη σειρά που σας ανέφερα, αν και δεν υπήρχε ε, λόγος που σας ανέφερα με αυτή τη σειρά. Ο Ευάγγελος, λοιπόν, πρώτα. Οι τεχνικοί θα ανάψουν το μικρόφωνο σου. Καλημέρα. Good morning. My name is Evangelos Kassos and I'm a high school Λέγομαι Ευάγγελος Κάσος και είμαι φοιτητής από την καρδίτσα της Ελλάδας. Ήθελα να ενημερώσω φίλους και οικογένεια για τις ευρωεκλογέ. Όλοι ήταν ενθουσιώδεις και πολλοί με ευχαρίστησαν. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι λόγω των διαδικασιών μπερδεύτηκαν και δεν ήξεραν που πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να δημιουργήσουν μια μικρή ομάδα που να ενημερώνει αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν και έτσι οι ψηφοφόροι δεν θα μπερδεύονται όταν πάνε στα εκλογικά κέντρα ή δεν θα βαριούνται και θα μπορούν να ε, βρουν το χρόνο για να πάνε ένα ποτό ε, μετά για να γιορτάσουν. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στη Μάλτα, είτε στην Αυστρία. Στην, ε, στο Δήμο τη Καρδίτσα οργανώσαμε τοπικέ εκδηλώσει που επικεντρώνονται στο να κάνουν τον κόσμο να κινητοποιηθεί, να ενημερωθεί για την εκλογική διαδικασία και τι λεπτομέρειε και για του ψηφοφόρου. Ε, η όλη δράση ήταν ε, πολύ επιτυχημένη και είχαμε τουλάχιστον 500 συμμετοχέ. Όταν λοιπόν αναρωτιέστε τι μπορώ να κάνω για να ε, ενεργοποιηθώ, το πρώτο είναι να δημιουργήσετε μια τέτοια ομάδα για τι εκλογέ, για να προσελκύσετε περισσότερου ψηφοφόρου. Είναι εύκολο να δημιουργήσει κανεί με τέτοια ομάδα. Πώ, πρώτο βήμα. Πρώτα απ' όλα διαλέξτε τουλάχιστον 5 άτομα για να ξεκινήσει ένα chat στο Facebook, στο Messenger, στο WhatsApp από όπου θέλετε. Μετά διαλέγετε κάποιον που είναι υπεύθυνο τη ομάδα, εσεί ο ίδιο προφανώ, που φροντίζετε όλοι αυτοί να γνωρίζουν πώ γίνονται εκλογέ, πώ ψηφίζει κανεί. Και πηγαίνετε στο European slash ε, elections EU για να ενημερώσετε. Μετά φροντίζετε να ε, στείλετε μηνύματα και βίντεο με το, χρησιμοποιώντα το hashtag ε, voting squad. τα βάζετε στο facebook και στο instagram και προσκαλείτε τουλάχιστον άλλου πέντε να κάνουν το ίδιο. Έτσι βλέπουμε αυτέ οι ομάδε να κάνουν πολύ καλή δουλειά και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ που παρέμεινε και στα δύο λεπτά. Αυτό ακριβώ είναι ο χρόνο ομιλία που πολλοί ευρωβουλευτέ, πολλά μέλη ε, λαμβάνουν όταν ε, μπορούν να τοποθετηθούν στο ημικύκλιο κατά τη συζήτηση. Δύο λεπτά ομιλία. Χαβιέρ, ποια είναι η δική σου πρόταση. Ευχαριστώ, με λένε Χαβιέ Ροντρίγκε και αυτό είναι το δικό μου πρόγραμμα δράσης για να προσελκύσω εγώ ψηφοφόρους. Λέγεται ε, ένα πιντσοπότε για την ε, Ευρώπη. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους μπάρμαν στην περιοχή μας του Σαν Σεμπαστιάν μια από τις πρωτεύουσε ε, της χώρας των Βάσκων που, έχω, που ζω εγώ στην Ισπανία και είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί κανείς να πάρει ένα πίντσο και ένα ποτό για μειωμένη τιμή. Ε, δηλαδή κάτι σαν μεζέ και ποτό στο happy hour, ε, συγκεκριμένη μέρα και ώρα της εβδομάδας. Είναι μια πρωτοβουλία που ε, την ξέρουν όλοι πια στην πόλη ε, και στην ευρύτερη περιοχή και ξέρουμε όλοι καλά τι θα πει πίτσο πότε, happy hour δηλαδή. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που μπορεί να συγκεντρώσει τον κόσμο για να αισθανθεί ευδιάθετο. Για να οργανώσει καλή λοιπόν ένα τέτοιο πιντσοπότε αρκούν τρία βήματα. Πρώτα απ' όλα να φροντίσει να έχει όλε τι προμήθειε. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει ως μεζέδες ό,τι είναι διαθέσιμο και ό,τι είναι πιο εύκολο. Δεύτερο βήμα είναι να βρει κανείς ένα μέρος όπου μπορεί να συγκεντρώσει όλο τον κόσμο που θέλει να συγκεντρώσει. Είναι πολλές οι επιλογές. Μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο χώρο ή στο σπίτι του κιόλα. Σε ένα ιδιωτικό χώρο ή και σε ένα χώρο όπω ένα μπαρ. Το επόμενο βήμα είναι να προωθήσει κανεί την εκδήλωση χρησιμοποιώντα το κοινωνικό του δίκτυο. Δηλαδή να ενημερώσει φίλου, οικογένεια και Τέλος, βεβαίω πρέπει αυτό να υλοποιηθεί. Ε, Αυτή είναι η εκδήλωση και βρίσκω ότι είναι το ωραιότερο περιβάλλον, ο ωραιότερο χώρο για να συγκεντρωθεί όλο αυτό ο κόσμο που μπορεί σε καλή διάθεση να πάρει τι πληροφορίε για τι εκλογέ, να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουν και τι δύναμη έχουν στα χέρια του με την ψήφο του. Αυτά ήταν τα πρώτα βήματα που εγώ μπορώ να σα προτείνω για να ε, υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα δράση. Στο καλό δεν χρειάζεται πάρα πολλά για να γίνει όλο αυτό. Αρκεί ε, να αρχίσει κανεί να δουλεύει και από το σπίτι. Ευχαριστώ. Και η τρίτη πρόταση φίλοι μου από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από ένα μήνα ήμουν εδώ στην πρώτη σύνοδο του Κοινοβουλίου για τους νέους και πήρα τον λόγο. Δεν είμαι από τα μεγαλύτερα κράτη της Ευρώπης και ήταν απίστευτο που για πρώτη φορά μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα μου σε μια ευρωπαϊκή ε, σύνοδο. Ε, στις εκδηλώσεις για τους νέους ουδέποτε ήταν ε, δυνατόν να μιλήσουμε ε, την μητρική μας γλώσσα όλοι από οποιοδήποτε κράτος. Σήμερα λοιπόν έχω προσκληθεί να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση που είναι μια φανταστική ευκαιρία για να εκφράσουμε την ευρωπαϊκή γλωσσική ποικιλομορφία και πολιτιστική ποικιλομορφία και η στιγμή για μένα είναι ιστορική. Είμαι λοιπόν πραγματικά πολύ χαρούμενος. Και τώρα ε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω όντως τη μετρική μου γλώσσα. Όπως βλέπετε λοιπόν Έγινε και η διακόσμηση με τα σύμβολα τα οποία γνωρίζετε ήδη. Και εμείς επιλέξαμε να πούμε το εξή. Ε, ως μήνυμα θα ψηφίσεις ναι ή όχι. Και πολλοί πέρασαν από την πόρτα του ναι. Κάποιοι απέφυγαν να περάσουν από τις δύο πόρτες αυτές για να διαλέξουν αν θα ψηφίζουν ή όχι. Έχουμε λοιπόν τέτοιες ε, ε πόρτες ε, στα σχολεία, στις πλατείες, σε δημόσιους χώρους όπου περνάει πολλοί κόσμος και κόσμος που ενδεχομένως να μην ξέρει τόσο πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διοργανώνουμε λοιπόν τέτοιες εκδηλώσεις για να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, αλλά τελικά η καλύτερη μέθοδος είναι η εξής, να πείσουμε τους νέους και να επηρεάσουμε αυτούς που δεν πέρασαν από καμία πόρτα. Δεν διάλεξαν μία πόρτα. Αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μένα και με την εκδήλωση αυτή κατάφερα να συναντήσω πολύ κόσμο που δεν είχα συναντήσει υπό άλλες συνθήκες. Και έτσι λοιπόν διοργανώνουμε ε, και εκδηλώσεις για τον τύπο, για τα μέσα ενημέρωσης. Μπορείτε να κοιτάξετε και τη σελίδα του κ. Κοβάτσκι στο facebook. Να ευχαριστήσω μεταξύ άλλων και τον ε, Ντάβιτ για την ε, βοήθεια που μας έδωσε. Σας ευχαριστούμε. So, here you go. Those were... Ε, αυτές ήταν οι τρεις προτάσεις λοιπόν για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εσάς. Τώρα αυτό που θέλω να σας ζητήσω είναι να μου πείτε αν έχετε ερωτήσεις για τους τρεις νικητές. Ερωτήσεις, κάποιο σχόλιο, μια αντίδραση. Θέλετε να τους ρωτήσετε τίποτα. Θέλετε να τους πείτε κάτι. Μπορείτε να λάβετε εσείς το λόγο. Και στη γλώσσα σας μάλιστα. Ποιος θέλει το λόγο, ποιος είναι αρκετά θαραλέος για να ανοίξει το χορό. Μια-δυο ερωτήσεις πρώτα και μετά θα απαντάει ο καθένας. Ναι, αν θέλετε να μιλήσετε παρακαλώ καλύτερα σταθείτε όρθιος και θα ξεκινήσει το μικρόφωνο. Πείτε μας και ποιοι είστε, συστηθείτε αν γίνεται, για να ξέρουμε και από πού είστε και ποιοι είστε. Δεν είναι ότι δεν μιλάω αγγλικά ή γαλλικά, αλλά θα μιλήσω τη μητρική μου. Είμαι η Ιωάννα από τη Ρουμανία και κέρδισα στο διαγωνισμό λοιπόν αυτό. Democracy and me. Δημοκρατία και εγώ. Και μίλησα λοιπόν για ένα λεπτό για το θέμα τη δημοκρατία και για το τι σημαίνει για μένα η δημοκρατία. Είχα λοιπόν μια ερώτηση να σα κάνω. Τα πράγματα είναι δύσκολα στη χώρα μου σε ό,τι αφορά τι εκλογέ. και δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε σε πολλέ περιπτώσει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θα μαζέψουμε και άλλε ερωτήσει. Ποιο θα ήθελε να κάνει κάποια άλλη ερώτηση ή να μας δώσει κάποια παρατηρήση να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιουλιάνα, από τη Γερμανία, 16 χρονών είμαι και είχα μία ερώτηση για το project για την εκδήλωση αυτή με τις ε, πόρτες ε, για ναι ή όχι. Μία ερώτηση. Τι κάνατε με τους ανθρώπους που πέρασαν από την πόρτα του όχι, ότι δεν θα ψηφίσουμε. Τους συζητήσατε για παράδειγμα γιατί δεν θα ψηφίσουν, πώς προσπαθήσατε για να του επηρεάσετε ενδεχομένω για να ψηφίσουν τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια ερώτηση. Mm. Ποιος θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση, ε, να κάνει κάποιο σχόλιο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ να ρωτήσω το εξή. Αν σε μία λέξη θα ήθελα να πούν γιατί, για ποιο λόγο να πάει να ψηφίσει κάποιος από 18 στο 80, ποια θα ήταν η κουβέντα αυτή, με ποια λέξη θα προσπαθούσαν να πείσουν. Μάλιστα και εγώ είμαι πολύ περίεργη. Άλλος ένας. Άλλη μια ερώτηση. Uh, το μικρόφωνο σας αν θέλετε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Από τη Ρουμανία είμαι, Βλαντιμίρη ονομάζομαι. Και εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση για την ομάδα αυτή. Τι θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους που δεν θέλουν να παναψηφίσουν. Okay, I uh, floor. Ευχαριστώ πολύ και να δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στους νικητές μας. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο να απαντάει, να απαντήσει. Έχουμε ένα λεπτό για τον καθένα και θα μας μείνει και χρόνος να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο για να ξεκινήσει τις απαντήσεις. Ένα λεπτάκι έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη ερώτηση της Γιωχάννα για το τι είναι πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τι εκλογές. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να ξυπνήσω το ενδιαφέρον του κόσμου για τις ε, εκλογές και μάλιστα σε ανθρώπους, σε πολίτες που δεν ε, ενδιαφέρονταν. Άρα δεν έχει μεγάλη σημασία να μιλάω για τις εκλογές με τους φίλους μου, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι δεν σκόπευαν να πάνε να Επίσης έγινε άλλη μια ερώτηση τι θα λέγαμε στον κόσμο που δεν πέρασε από την πόρτα του ναι. παρακαλήσαμε τον πολίτες να μας πούν γιατί δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν και να το κάνουν και γραπτά. Και αν ε, θα διάλεγα μία λέξη, ένα σλόγγαν ε, για τις εκλογές, θα έλεγα ότι οι εκλογές είναι σεξι. Και να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί είναι σεξι. Και τελευταία ερώτηση Καλή ιδέα θα τον θεωρώ να παρατρένουμε τον κόσμο να βγει στον δρόμο, να διαδηλώσει, να δημιουργήσει ένα κόμμα για κάπως να προωθήσει τις ιδέες του, εν πάση περιπτώσει. So, who of you two will take over? Μάλιστα, λοιπόν. Ποιος θα πάρει το λόγο? Okay, so uh, I will answer in Spanish, so the ones that don't speak Spanish, please. Θα μιλήσω ισπανικά, γι' αυτό παρακαλώ όσοι δεν μιλάτε ισπανικά, βάλτε ακουστικά. Ε, la primera pregunta. Πρώτη ερώτηση. που θέσατε εσείς από τη Ρωμανία είναι πως ε, ε, βρίσκουμε κίνητρα ώστε ε, ο κόσμος και κυρίως οι νέοι να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχάς πιστεύω πως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ότι στην ουσία έχουν ένα είδος εξουσίας, ότι από εκείνους εξαρτάται λοιπόν, να αποφασίσουν ποια μορφή θα έχει η μελλοντική κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πάει κανείς να ψηφίσει και ότι τελικά είναι κομμάτι μιας διαδικασίας μέσω της οποίας η κοινωνία ε, συμφωνεί ή όχι, διαφωνεί με το πώς θα χαράξει το μέλλον της. Έπειτα, τι θα έλεγα με μια λέξη, ε, η λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι η λέξη δημοκρατία. Και έπειτα, τι θα έλεγα στους παππούδες μου ή στους πιο ηλικιωμένους που δεν πάνε να ψηφίσουν ε, για οποιοδήποτε λόγο. Θα τους έλεγα ότι όπως... Ε, η γιαγιά μου με φροντίζει, μου φτιάχνει φαγητό και με ή απλά και μόνο ανησυχεί για μένα ότι θα πρέπει να ανησυχεί και για μένα και με το να πάει να ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ευάγγελος. Και εγώ θέλω να μιλήσω στα ελληνικά, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Ε, καταρχάς, ε, θα ήθελα να συνδυάσω τις δύο ερωτήσεις, το πώς θα ενθαρρύνουμε τους ψηφοφόρους, τους νέους ψηφοφόρους και τι γίνεται με τους ηλικιωμένους ανθρώπους και πιστεύω ότι εδώ είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μέσα από έρευνες που έχουν γίνει οι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό το οποίο βγαίνει και πάει να ψηφίσει δεν, οι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτό το σύστημα της δημοκρατίας. έχει γίνει μέρος της ζωής τους, οπότε δεν νιώθουν ε, την ανάγκη να μην πάνε να ψηφίσουν. Το θεωρούν, ε, ε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που η ψήφος είναι και υποχρεωτική, ε, το θεωρούν υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουν και, και η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Τώρα, ε, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε στους νέους ανθρώπους είναι ότι οι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ε, πηγαίνουν να ψηφίσουν. Θα αφήνατε ποτέ τους ηλικιωμένους, τη γιαγιά σας ή τον παππού σας να, ελέγξει, να, να καθορίζει το τι θα ανεβάζετε στο facebook, στο instagram ή το, τι θα, ή το τι θα φορέσετε για να βγείτε έξω. Όχι. Οπότε γιατί αφήνετε τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους γονείς σας, τους, ε, τους ε, παππούδες σας, τις γιαγιάδες σας να πάρουν πολύ σημαντικότερες αποφάσεις για το μέλλον σας. Οπότε θα ήθελα και έτσι σαν μια λέξη να περιγράψω τις εκλογές με τη λέξη μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. So, thank you for this, ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ καλή αυτή επικοινωνία και το γύρο ερωταπαντήσεων. Σας, τώρα το μπαλάκι είναι δικό σας, στο γήπεδό σας. Να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε ένα κωδικό στην, στο μηχάνημα ψηφοφορίας μπροστά σας. Κοιτάξτε και το σλάιντο, βάλτε το στο Google αν θέλετε, πάτε στην ε, κεντρική σελίδα και βάλτε τον κωδικό αυτό. Εκεί που σας ζητάει τον κωδικό. Και θα μπείτε λοιπόν ε, ε, μια σελίδα που έχουμε δημιουργήσει για τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση. And what I would now like to ask you is to... Και τώρα λοιπόν αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι να σκεφτείτε λίγο ο καθένας τον εαυτό του τι θα πρότεινε να κάνει για να καλέσει τους φίλους του, τους γείτονε του, να τους παροτρύνει να πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Πώς μπορούμε λοιπόν να παρατρένουμε φίλους και γείτονες να ψηφίσουν. Έχετε δύο λεπτάκια. Γράψτε μας αν θέλετε την πρότασή σας, μία ή και πιο πολλές. Τι θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε εσείς προσωπικά για να παρατρύνετε τον κόσμο να ψηφίσει. It's great, you're productive. I already have 10 ideas.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 ideas are still 100. <laughs> Um, Φτάσαμε τους 100. Λοιπόν, ωραία. Σίγουρα αν σας αφήνω ένα πεντάλεπτο θα συμπλήρωναν κι άλλοι. Αλλά Αντί να κοιτάει ο καθένα μόνο στο το τηλέφωνό του, θα ήθελα να γυρίσετε στο γείτονά σα προ τα αριστερά, όσες, όσοι έχετε κάποιο γείτονα προ τα αριστερά, κάπω θα τα καταφέρετε. Και έχετε τέσσερα λεπτά σε ζεύγη, τέλο πάντων σε δίδυμο, να εκθέσετε την ιδέα σας ο ένας τον άλλο, την καλύτερη που σας ήρθε, δύο λεπτά για τον ένα και δύο για τον άλλο και θα σας κάνω εγώ νόημα στο δίλεπτο για να αλλάξετε μεταξύ σας. Like to, uh, do is discuss... Θέλω λοιπόν να συζητήσετε με τον γειτονά σας τη δική σας ιδέα πρώτα και να πείτε γιατί πιστεύετε ότι θα πετύχει και ότι θα πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Θα αρχίσει να γίνεται λίγο φασαρία τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Βρήκατε όλοι κάποιο γείτονα για να συζητήσετε. Πάμε.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 20 more seconds to go. Okay. Okay, time's up. Τέλειωσε ο χρόνος. έγινε και λίγη, λίγος τζερτζελέ στο κοινοβούλιο. Τώρα να ακούσουμε μερικές από αυτές τις ιδέες, αλλά όχι από αυτόν που τη σκέφτηκε. Θέλω ο γείτονα να μας εξηγήσει την ιδέα που άκουσε, εάν ήταν κάτι πολύ πιστικό και κάποια ιδέα ήταν πολύ καλή. αν ήταν κάτι που θεωρεί πολύ πετυχημένο, πολύ αποτελεσματικό. Και πάλι λοιπόν χρόνο για να παρουσιάσουμε την ιδέα του γείτονα. Ποιο θέλει να κάνει την παρουσίαση, εδώ, στην πρώτη σειρά έχουμε μία. Καλημέρα, είμαι από την Αταλία και είμαι από την ε, Λετωνία. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν την ε, μετρική μου γλώσσα. Ο γείτονά μου είχε την ιδέα να προσφέρει τρόφιμα. Φαΐ στον κόσμο ή τέλο πάντων κάποιο πρωινό να φάνε όλοι μαζί κάτι τέτοιο. Εγώ βρίσκω ότι θα μπορούσε να πετύχει κάτι τέτοιο. Thank you. Yes, please. My name is Asha and I'm from Finland. Uh... Με λένε Άσα από τη Φινλανδία. Η γείτονα μου η Βέρα είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Uh, Είπε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε βίντεο που να εξηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα βάζουμε στο YouTube. Να λένε τα βίντεο τι κάνουν για μα, τι κάνει για μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί περισσότεροι δεν ξέρουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μα. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Να εξηγήσουμε τι, κάνουν, ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μα. Ένα χειροκρότημα για όλε αυτέ τι ιδέε. Να και μια άλλη. Για να πάμε από εκεί. Γεια σα. Είμαι η Κριστίνα από την Ισπανία και θα μιλήσω Ισπανικά. Ο vecino ha tenido una muy buena ε, Ο γειτονά μου είναι από τη Σλοβακία και μου είπε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να, να να καθίσουμε όλοι μαζί στην οικογένεια και κάποτε στη Σλοβακία οι παλιότεροι δεν μπορούσαν καν να ψηφίσουν. Το ίδιο συνέβαινε και στη δική μου χώρα όπου είχαμε δικτατορία για πάρα πολλά χρόνια ε, και όταν κανείς δεν είχε την ευκαιρία να ε, ψηφίσει ενώ τώρα πια έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει θα έπρεπε να το κάνει, να του τιμήσουμε τα παλιά. Ναι, παρακαλώ. Και εγώ θα μιλήσω στα, στη γλώσσα μου. Um Εμεί είχαμε μια άλλη ιδέα. Αν ε, καλούσαμε κόσμο να μιλήσει για, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάναμε παλιότερα σε αυτές τις διάφορες εκδηλώσεις για τους νέους, έρχεται κόσμος, αλλά έρχεται ο κόσμος που ήδη ενδιαφέρεται δεν αρκεί αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε τον κόσμο που δεν ενδιαφέρεται να ενημερωθεί. Το βλέπουμε και στα σχολεία ότι οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται, παιδιά που δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν πάνε καν να ψηφίσουν, άρα γιατί να έρθουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν γι' αυτό η ιδέα με τις πόρτες είναι ενδιαφέρουσα γιατί εκεί υπάρχει μια επαφή αλλά και αντιπαράθεση. Ο κόσμος δηλαδή πρέπει να πει και να εξηγήσει γιατί ε, κρατάει αυτή τη στάση. Αυτή η... Αυτό επιτρέπει στον κόσμο να πει <clears throat> ναι, εγώ δεν θέλω να πάω να ψηφίσω γιατί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μου είναι αδιάφορη, δεν νοιάζει τι γίνεται, είναι πολύ μακριά από την καθημερινότητά μου. Αν καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει κοντά και να μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έρθουν μόνο οι ε, ε, ενδιαφερόμενοι ήδη, ενώ θα μπορέσαμε να προσελκύσουμε και αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Μάλιστα, βλέπω και άλλους. Δύο εκεί πίσω-πίσω. Και εδώ... Εντάξει, αρχίσουμε εκεί πίσω-πίσω και θα δούμε με πόσο χρόνο έχουμε ακόμα για να μιλήσουμε. Ναι, ε, εσείς. Δεν ακούγεται η ομιλήτρια, δεν έχει μικρόφωνο. Ναι, γεια σας. Τα ξαναλέω από την αρχή. Λοιπόν, γεια σας, εγώ είμαι από τη Λετωνία. Η γειτόνισσα μου είχε την ιδέα να δώσουμε ένα μικρό δωράκι σε κάποιον ε, που πάει να ψηφίζει για πρώτη φορά. Ήταν μια μικρή καρτούλα, ένα μικρό κέρμα, νόμισμα, ενθύμιο ή ένα γλυκάκι, σαν να ήταν ε, τη γενέθλια. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν κανείς ψηφίζει για πρώτη φορά. Ε, να το γιορτάσουμε με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ναι, και εσείς στην προηγούμενη σειρά. Μισό, λεπτό, κάποιο ακόμα είχε ε, ζητήσει το λόγο. Ναι, όχι, εσεί, εσεί. Sorry, very, uh, my name is Emilia and I am... Εγώ ονομάζομαι Εμίλια και είμαι από τη Λιθουανία. Και θα ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου. Ε, γείτονά μου πρότεινε κάτι πολύ καλό, να μιλήσουμε για το παράδειγμα του Brexit. Το πώς δηλαδή όταν οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν, τι μπορεί να συμβεί. Ότι η ψήφος των νέων έχει μεγάλη επιρροή και οι νέοι δεν πρέπει να φοβούνται να ψηφίσουν και να πούν τη γνώμη τους σε εθνικό επίπεδο. Uh, Τρεις. Τρεις ακόμα θα ακούσουμε και μετά θα κλείσουμε γιατί θα ξεκινήσει η επόμενη συνεδρίαση. Ε, η κοπέλα με το κόκκινο. Ευχαριστώ. Εγώ ονομάζομαι Σαρλότ, είμαι από τη Γαλλία και θα μιλήσω γαλλικά. Ε, εμένα με ενοχλεί κάτι αρκετά έντονα σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων στις ευρωεκλογέ και σε σχέση με γενικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε με τους νέους, στη Γαλλία τουλάχιστον, οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν καν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το πολύ αφηρημένο. Δεν συνειδητοποιούν τι γίνεται και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ με την εταιρεία και την οργάνωση με την οποία είμαι εδώ έχω κάνει ένα project ε, για να μιλήσουμε για τη συμμετοχική δημοκρατία με τους νέους, για να σκεφτούμε νομοθεσίες, νομοθετήματα για το μέλλον που θέλουμε να φτιάξουμε. Δηλαδή να μην λέμε μόνο αν δεν πηγαίνετε να ψηφίσετε γιατί οι ευρωεκλογές είναι σεξι, αλλά γιατί Υπάρχουν ιδέες, ε, προσπαθήστε να στηρίξετε αυτά που σας ενδιαφέρουν και προσπαθήστε να αλλάξετε τα, πράγματα, τα πράγματα με τις ιδέες σας και όχι μόνο να δέχεστε ιδέες που σας έρχονται ούρανο κατέβετες και που δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνουν. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Τώρα είναι το δυνηρό κομμάτι. Ποιον, να διαλέξω queuing Εσείς εδώ περιμένετε αρκετή ώρα. Το νέο... Εσείς εδώ και μετά ο νέος με το μπλε. Hello, Ονομάζομαι Λούκα, είμαι από τη Γερμανία, είμαι 18 χρονών και θα μιλήσω ρουμανικά. Πιστεύω πως είναι μια καλή ιδέα να σκεφτούμε τα σχολεία ε, και να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στη Ρουμανία δεν είμαστε πολύ οργανωμένοι. Πρέπει κανείς να καταλάβει πώς δουλεύουν οι ευρωεκλογέ και τι σημαίνουν. Όχι μόνο στη Ρουμανία. Πολλοί νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν ξέρουν καν τι, ποιο είναι το ζήτημα. Να εξηγήσουμε στους νέους πώς, τι σημαίνει, να τους δώσουμε το κίνητρο, να τους ενθαρρύνουμε να πάνε να ψηφίσουν γιατί οι εκλογές βοηθάνε στο να συμμετήσουμε το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Εσείς τώρα. Εγώ είμαι από την Ισπανία και θα μιλήσω ισπανικά. επειδή είναι δύσκολη και πολύ σοβαρή η κατάσταση με τις ευρωεκλογέ. νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε στους νέους την ιδέα ότι όλα αυτά μπορούν να είναι και διασκεδαστικά πέρα από τη σοβαρότητα του θέματος και εδώ με τις γειτόνισσές μου μιλήσαμε για κάτι διασκεδαστικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τους νέους αποφασίσαμε να μοιράσουμε προφυλακτικά στους νέους με το σύνθημα «Μα είναι η πρώτη σου φορά» γιατί παρόντος πολλοί νέοι πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά και είναι μια ξεκάθαρη ιδέα και ε, που μπορεί να μείνει στο μυαλό τους με ένα προφυλακτικό που λέει είναι η πρώτη σου φορά. <laughs> Το τελευταίο ήταν καλό ε, πρέπει να πω. Όμως ο χρόνος ε, πετά και δυστυχώ δεν μπορώ να ακούσω άλλου άλλους που θα μου πούνε τι είπαν οι γείτονε. Αλλά μετά στο διάλειμμα σα καλώ να το κάνετε, να συζητήσετε και να σκεφτείτε όλα αυτά γιατί πραγματικά από εμά εξαρτάται να δώσουμε και να, κίνητρα και να παροτρύνουμε τους άλλους. Γιατί εμείς είμαστε υπεπισμένοι όπω είπατε πολλοί από εσά, αλλά πώ μπορούμε να πείσουμε και του υπόλοιπου. Τελευταίο στοιχείο, πριν να δώσω το λόγο και να ξεκινήσει η επόμενη συνεδρία, θα ήθελα να σας ζητήσω να χρησιμοποιήσετε το, το άλλη μια φορά και να απαντήσετε σε, στο εξή. Αυτή τη φορά ψηφίζω. Ε, αυτό δεν είναι μόνο ένα σύνθημα για να καλέσουμε άλλους να ψηφίσουν και εκείνοι. Είναι και η ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε για τι πράγμα ψηφίζουμε, για ποιο λόγο ψηφίζουμε. Ένα-δύο λόγια λοιπόν για το γιατί ψηφίζετε εσείς οι ίδιοι. looks good. big overview. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ε, των ε, αξιών που έχουμε όλοι μας ε, και γι' αυτό ψηφίζουμε. Και ελπίζω αυτό να ψηφίσετε και εσείς. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας για αυτή την ε, πρώτη αυτή ε, ε, εκδήλωση, το πρώτο αυτό πάνελ. ευχαριστήσουμε και τις ερμηνείς για την ερμηνεία. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Κριστόφ για να διοργανώσει το δεύτερο πάνελ.